Προχωρούμε τώρα στις ψηφοφορίες. Έκθεση Αρτουή. Ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται έκθεση Κάσπαρη. Ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση Ουιχέη. Ψηφοφορία με ονομαστική κλήση Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση Άντερσον. Τροπολογία αριθμός 96 με ανάταση της χειρός. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 95 ψηφοφορία με ονομαστική κλίση αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Η τροπολογία 95 είναι σε διάρκεια ψηφοφορίας. Ψηφοφορία με ονομαστική κλίση τελείωσε η ψηφοφορία. Από ό,τι μου λένε υπήρξε κάποιο πρόβλημα με τη διερμηνία. Θα επαναλάβουμε την ψηφοφορία, παρακαλώ χωρίς φωνές. Επειδή υπήρξε κάποιο πρόβλημα με τη διερμηνία, θα επαναλάβουμε την ψηφοφορία στην τροπολογία αριθμός 95. Ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Αρχίζει ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. εγκρίνεται που σημαίνει ότι η πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περατώθηκε. Έκθεση Λούντγκρεν, τροπολογία 41, ψηφοφορία μονομαστική κλίση, αρχίζει ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. εγκρίνεται που σημαίνει ότι η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου περατώθηκε. Έκθεση Γκροστέτ. Το επόμενο θέμα είναι η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας για την έναρξη διαπραγματεύσεων βάσει της έκθεσης της κυρίας Γκροστέτ για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας Επιθυμεί κανείς να μιλήσει υπέρ της απόφασης της Επιτροπής για την έναρξη διαπραγματεύσεων. Δεν βλέπω. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπούτι Κόφερ για να μιλήσει κατά της απόφασης της Επιτροπής για δύο λεπτά. Κύριε Μπούτι Κόφερ, έχετε το λόγο. Thank you, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λακωνικότατα. Πιστεύουμε ότι πρέπει να ληφθεί εδώ αυτή η απόφαση έχει μεγάλη σημασία για την ε, κοινή μας δουλειά και ύπαρξη. Είμαστε υπέρ της κοινή ανάπτυξης κοινών δραστηριοτήτων από όλους εμάς τους Ευρωπαίους για την κοινή μας ασφάλεια. Και αυτό σημαίνει συνεργασία στο χώρο και της βιομηχανίας της ασφάλειας. Ωστόσο εδώ έχουμε να κάνουμε με μια χαμένη ευκαιρία. Αυτό βλέπουμε εδώ. 178 διαφορετικά οπλικά συστήματα που έχει η Ευρώπη δεν πρόκειται να μειωθούν, δεν θα μειωθούν οι κατάλογοι των προμηθειών, δεν θα εξοικονομήσουμε πόρους. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα επιτευχθούν συνολικά οι στόχοι που έχουν προαναγγελθεί. Γι' αυτό δεν θέλουμε αυτή την πρόταση. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα για την ασφάλεια. Χρειαζόμαστε περισσότερη αποτελεσματικότητα, οικονομία σε ε, εξαγωγική βιομηχανία ασφάλειας και εξοπλισμών. Κατά της απόφασης Επιτροπής ζήτησε το λόγο η κυρία Γκροστέτ για δύο λεπτά να μιλήσει υπέρ της απόφασης Επιτροπής. Κυρία Γκροστέτ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Στις 21 Φεβρουαρίου του 2017 η Επιτροπή ΙΤΡΕ με μεγάλη πλειοψηφία ενέκρινε την έκθεσή μου για το, για το βιομηχανικό πρόγραμμα άμυνας καθώς και την διαπραγματευτική εντολή. Σας ζητώ λοιπόν να στηρίξετε επιβεβαιώνοντας σήμερα την λιμένη απόφαση της Επιτροπής ΙΤΡΕ για να ξεκινήσουμε τις διοργανικές διαπραγματεύσεις. Ο κανονισμός αυτός ε, στόχο έχει την ε, υποστήριξη της ε, βιομηχανικής συνεργασίας στην Ευρώπη ώστε να καταστήσουμε πιο ανταγωνιστική την βιομηχανία μας και να δώσουμε κίνητρα για την καινοτομία. Θέλουμε να αναπτύξουμε την βιομηχανική και τεχνολογική βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφεύγοντας τις περιτές και δαπανηρές επικαλύψεις. Οι συμπολίτε μας απαιτούν από μας να δράσουμε υπέρ της ασφάλειάς τους. Ήρθε η ώρα να βελτιώσουμε τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από αστάθεια. Ο κανονισμό αυτό θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ την 1η Πρώτου του 2019. Θα πρέπει λοιπόν το συντομότερο δυνατό να το θέσουμε σε ισχύ και να τον εγγράψουμε στον προπολογισμό του 2019. Γι' αυτό σα παρακαλώ να στηρίξετε την απόφαση, να υπερψηφίσετε την πρόταση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ. Ακούστηκαν και οι δύο προτάσεις. Θέτω την απόφαση της Επιτροπής σε ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η πρόταση της Επιτροπής που σημαίνει ότι η Επιτροπή μπορεί να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με άμεση ισχύ. Προχωρούμε στην έκθεση Φορέντσα Μπιόρκ, παράγραφος 14 του αρχικού κειμένου με ανάταση της χειρός. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θέλετε να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Ωραία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την παράγραφο 14. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λήξη ψηφοφορίας εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Αιτιολογική σκέψη LA του αρχικού κειμένου υπέρ κατά αποχές θα κάνουμε εδώ ηλεκτρονικό έλεγχο αρχίζει ψηφοφορία λήξη ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Αιτιολογική σκέψη LA του αρχικού κειμένου υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Θέλετε τσεκ. Θα κάνουμε και σε αυτό ηλεκτρονικό έλεγχο. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λήξη ψηφοφορίας εγκρίθηκε με καθαρή πλειοψηφία. Ψηφοφορία με ονομαστική κλίση για το σύνολο του κειμένου. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λήξη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Προχωρούμε στην έκθεση Τζουφρίντα για το σύνολο του κειμένου ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Αρχίζει η ψηφοφορία. λήξη ψηφοφορίας εγκρίνεται και προχωρούμε στην έκθεση Βαλίνα τροπολογία 1 στην παράγραφο 4 από 76 και παραπάνω μέλη του Κοινοβουλίου ψηφοφορία με ονομαστική κλίση αρχίζει η ψηφοφορία. Λήξη ψηφοφορίας απορρίπτεται. ψηφοφορία με ονομαστική κλίση για το σύνολο του κειμένου αρχίζει η ψηφοφορία. λήξη ψηφοφορίας εγκρίνεται ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες σας ευχαριστώ πολύ. Προχωρούμε τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις αιτιολογήσεις ψήφου. Ξεκινούμε με την έκθεση του κυρίου Ουιχέλη. Το λόγο έχει ζητήσει